Η Sitzung ist eröffnet. Συνόδου, αρχίζει συνεδρίαση. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Αν σας ενοχλώ κυρίες και κύριοι, να μου το πείτε. Ansonsten würde ich Sie bitten, Platz zu nehmen. σας παρακαλώ να καθίσετε. Vielen Σας ευχαριστώ. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κώδικα για τα μέλη των ε, Ευρωβουλευτών σε ό,τι αφορά τα οικονομικά συμφέροντα και τη σύγκρουση των συμφερόντων, χθες, 15 Ιουλίου 2014, σχετικά με τα πέντε μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ε, τα ονόματα